ένα πράγμα που λέγεται... Συντώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Ήμουν σε συνάντηση που άργησε να τελειώσει. Ε, δεν το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς ξέχασα και τα γυαλιά μου στην αίθουσα εκείνη. Θα δούμε αν θα τα καταφέρω τώρα χωρίς τα γυαλιά μου. Βλέπω ωστόσο ότι δεν δείχνεται κανένα ήκτο. Ε, για μένα ε, ζητώ ε, συγγνώμη και πάλι και ιδίω απέναντί σας σε εσά που ήρθατε έγκαιρα. Πρόκειται για το θέμα για το blockchain. Θα ακούσουμε παρουσίαση για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τις πολιτικές ε, αναφορικά με τα blockchain. Η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών είναι συνδεδεμένη επιτροπή υπό την ισχύ του άρθρου 54 και έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο συνήθως. Δηλαδή για ζητήματα προστασίας και επιβολής του νόμου. Υπάρχει τώρα μια επιτροπή η οποία συναπαρτίζεται από μέλη διαφόρων επιτροπών, intercommittee δηλαδή, αλλά θα σας τα πει καλύτερα η κυρία Γκόμες. Έχετε το λόγο, Άννα για το ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό θέμα. Θα ακούσουμε τις προτάσεις σας για το blockchain. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως είπατε, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για έκθεση που συντάσσεται για λογαριασμό της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, δηλαδή απευθύνεται σε αυτήν εφόσον είναι γνωμοδότηση, διότι το blockchain είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει, διευκολύνει τις εμπορικές ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επίσης ως σκοπό να ενισχύσει την εμπορική μας πολιτική, να διευκολύνει τις κινήσεις των τελωνίων, το εμπόριο γενικότερα. Επίσης, να εγγυηθεί την ασφάλεια σε διαμεθοριακές συναλλαγές, Εμείς τονίζουμε ότι πρόκειται για τεχνολογία η οποία θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη στις διάφορες ε, συναλλακτικές δραστηριότητες που εξαρτώνται βέβαια από τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις σχετικές συναλλαγές. δεν αναπτύσσει τη τεχνολογία αυτή μόνο από πολυεθνικές, ενδιαφέρονται και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θα πρέπει και αυτές να ωφεληθούν από τα ωφέλη που προσφέρει το blockchain. Αυτή ωστόσο η εικόνα είναι υπερβολικά ρόδινη. για κάτι που είναι σχεδόν απόκριφη επιστήμη αυτή η τεχνολογία blockchain. Εγώ μπορώ να φανταστώ ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί όντω να προσφέρει ισχύ και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για κακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι η τεχνολογία blockchain ξεκίνησε από τα κρυπτονομίσματα και όλο και περισσότερο πιστεύω θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και ε, να είμαστε ενήμεροι για το τι σημαίνουν αυτά τα κρυπτονομίσματα. Και να αναρωτηθούμε και με ποιον τρόπο μπορεί να προάγεται το δημόσιο συμφέρον, το κοινό συμφέρον δηλαδή και το δημόσιο συμφέρον με την τεχνολογία αυτή, διότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει και εγκληματικά συμφέροντα σε ε, ε, προσπάθειες ε, νομοποίησης παράνομων εσόδων. Όπως είπατε υπάρχει βεβαίως και το άλλο θέμα της προστασίας δεδομένων και της προσωπικής σφαίρας των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, που είναι βέβαια κρίσιμη σημασία αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Και είναι κάτι επίσης που ο εισηγητής το αναγνωρίζει, δηλαδή λέει ότι όντως υφίστανται προκλήσεις σχετικά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι και παραπάνω από προκλήσεις, πρόκειται για πραγματικές συγκρούσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι όντω σημαντικό που η παρέμβαση της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών θα επαναφέρει κάπως την πραγματικότητα αυτή την υπερβολικά αισιόδοξη ε, οπτική για κάποια πλονίκτηματα ασφαλώ μπορεί να υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται να δοθεί μια συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θεωρώ και συμφωνώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξει μια συμβουλευτική ομάδα blockchain για τις προδιαγραφές και τα πρότυπα και τα μέτρα που πρέπει να λεφθούν. Αυτή η συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται και από ειδικού της ασφάλειας ιδίως ό,τι αφορά την νομοποίηση παρανομεσόδων και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, αλλά και για τον κανονισμό GDPR, προστασία προσωπικών δεδομένων, όπου ε, μπορεί να προκύψουν ε, κίνδυνοι από την χρήση της τεχνολογίας blockchain. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στη συζήτηση τώρα. Η κυρία Μετσόλα πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Άννα Γκόμες, η συγγήτρια που παρουσίασε το σχέδιο εκθέσεως για το blockchain και εξήγησε πώς μπορεί να ενισχύσει την εμπορική πολιτική της Ένωσης η τεχνολογία blockchain που είναι και το επαναστατικό εκείνο στοιχείο που βλέπουμε σήμερα με τεράστιο δυναμικό ε, στη, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην φροντίδα της υγείας, στην ε, διαχείριση των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Βασικός μας στόχος εδώ πρέπει να είναι να δούμε πώς θα κρατήσουμε τα ωφέλη ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας τις εγγύησεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να υπάρχει ε, δεδομένη εμπιστοσύνη. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση και εντοπισμό των κινδύνων. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούν να μετριαστούν οι κίνδυνοι αυτοί ενώ ταυτόχρονα να επιτρέψουμε να αναπτυχθεί το δυναμικό του blockchain. Η εξέβρεση ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι σημαντική υπόθεση και πρέπει να δοθεί η αναγκαία νομική ασφάλεια στις ε, επιχειρήσεις για να μπορούν να επενδύσουν στη τεχνολογία αυτή με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων εγγύσεων, ιδίως απέναντι στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτή τη τεχνολογία ε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί κυρίως. Στην γνωμοδότηση δεν είμαι βεβαίω τεχνικός εμπειρογνώμων. Νομίζω όμως ότι το blockchain δεν αποθηκεύει παραδοσιακά δεδομένα, ώστε η τεχνολογία αυτή είναι συμπληρωματική των παραδοσιακών τραπεζών δεδομένων. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν μιλούμε για τους κινδύνους για την προστασία δεδομένων. Και ναι, μεν η τεχνολογία blockchain όταν ε, αποθηκευτεί κάτι εκεί μπορεί να το διαβάσουν πολλοί, αλλά όχι με ευανάγνωστο τρόπο. Υπάρχει και το ε, θέμα των κρυπτονομισμάτων, όπου συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να δούμε εκεί και τους κινδύνους του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την ε, τεχνολογία blockchain. Βεβαίω θα συνεργαστώ με όλες και όλους τους συναδέλφους για να εξασφαλίσουμε ότι το νομοθετικό μας σύστημα θα είναι τελικώς επαρκές και ισχυρό. Ευχαριστώ, Ρομπέρτα. Ντάνιελ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να διευκρινίσουμε το αντικείμενο της συζήτησης. Η πρόταση αυτή από την Επιτροπή Εμπορίου μιλάει για ιδιωτικέ εκδόσεις blockchain. Δεν αναφέρεται σε θέματα <clears throat> ε, κοινών ή δημοσίου τύπου εκδόσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των ε, δεδομένων, των τραπεζών δεδομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις κτλ. Και το θέμα είναι αν μπορούμε την τεχνολογία αυτή να την χρησιμοποιήσουμε στο διεθνές εμπόριο έτσι ώστε να ε, μειώσουμε τις, τα εμπόδια, τις τροχοπέδες που μπορεί να υπάρχουν ε, σε επίπεδο ελέγχων στις εξαγωγές-εισαγωγές. Πέρα από τον σκεπτικισμό ε, ορισμένων συναδέλφων είτε για τα blockchain είτε για τα κρυπτονομίσματα που δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Τα blockchain έχουν την δυνατότητα να επιτρέψουν ε, τα εμπορεύματα και το χρήμα να κυκλοφορεί χωρίς εμπόδια. Εγώ λοιπόν θέλω να αντιμετωπίσουμε σοβαρά λίγο τα θέματα αυτά αλλά να δούμε ακριβώς ότι τα blockchain δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά σε σχέση με την αποθήκευση δεδομένων. Από την άλλη υπάρχει θέμα σε σχέση ε, με, ε, την, με τις συναλλαγές. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται και δεν μπορεί να αποκριβεί. Συνεπώς λοιπόν στην παρούσα οικονομία σε σχέση ε, με την συναλλαγή σε ε, ρευστό φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο επώνυμο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να είμαστε σχετικά θετικοί λοιπόν για την δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας blockchain και πρέπει να είμαστε θετικοί και αυτό να φαίνεται στην έκθεση γιατί να δούμε πραγματικά ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα κρυπτονομίσματα. Η έννοια που λέει ότι, η λογική μάλλον, που λέει ότι η χρήση των κρυπτονομισμάτων είναι παράνομη είναι εντελώς λάθος. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή που να σχολιάσει τα, τις τροπολογίες, τις προτάσεις για τα blockchain. να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας στη γνωμοδότηση. Αυτά τα οποία είπατε θα ληφθούν υπόψη και από την Κοινή Επιτροπή και από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τίποτα άλλο. Δεν έχει λοιπόν ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει σε σχέση με την υπόθεση των blockchain. Οι Αμερικανοί περιμένουν βέβαια από πλευράς μας και από τέτοιες συναντήσεις να εκφραστούν οι απόψεις μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τις συζητήσεις μας και περιμένουν με ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα ακουστούν. Πάντως ευχαριστώ τα μέλη τα οποία είναι παρόντα εδώ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες και καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε αν κάποιες από τις τροπολογίες αυτές θα μπορούσαν να σχολιαστούν από, από πλευράς μας. Δεν ξέρω αν το ότι έχω κάποιες αμφιβολίες οφείλεται στην άγνοιά μου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα blockchain. και σε σχέση με το κατά πόσο διευκολύνουν την επωνυμία των συναλλαγών γιατί όχι αλλά μπορεί να υπάρξει και κατάχρηση αυτών των μέσων πληρωμών. Και μιας και δεν μιλάμε για ένα δημόσιο οργανισμό, αλλά για ιδιωτικού τύπου ε, εκδόσεις blockchain, αυτός δεν είναι λόγος, δεν συνιστά λόγο, εν πάση περιπτώσει, της μείωσης των ελέγχων και της αγνόησης των κινδύνων τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και σε σχέση και με την προστασία των ανθρωπίνων, των θεμελιωδών συγγνώμη, δικαιωμάτων. Κάποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από ορισμένε επιχειρήσεις και γι' αυτό ακριβώς αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει σαφώς να εφαρμόζεται το GDPR. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η πιο σημαντική συνεισφορά την οποία μπορούμε να δώσουμε εμείς μέσα από την γνωμοδότησή μας είναι για να διασφαλίσουμε το ότι αυτή η συμβουλευτική ομάδα η οποία θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες και για, την, για το βρώμικο χρήμα και για τα GDPR. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρώτη συζήτηση. Περιμένουμε με αγωνία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. έκθεση του ΩΣΑ για θέματα μετανάστευσης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Ζων Κριστόφ Ντεμό που είναι συντονιστής της ετήσιας έκθεσης του ΟΣΑ για τη μετανάστευση για το 2018 και για τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της μετανάστευσης στις χώρες του ΩΣΑ. Σας καλωσορίζουμε κύριε Τιμόν. Νομίζω ότι εξετάζοντας την έκθεσή σας έχουμε την δυνατότητα να συγκρίνουμε και να αντιπαραθέσουμε τις πολιτικές μας με άλλες περιοχές του κόσμου, του δυτικού κόσμου. Μπορεί επίσης να μας δώσει και ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε ε, να στεφθούν από επιτυχία. Και επίσης περιλαμβάνονται στοιχεία σε διάφορες χώρες ε, για την επίπτωση της μετανάστευσης στις αγορές εργασίας και περιλαμβάνει επίσης και επιμέρους σημειώσεις αναχώρα όπως επίσης και στατιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα για θέματα διεθνούς μετανάστευσης. Θα κάνετε λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση, συγγνώμη είναι πέμπτη απόγευμα μετά από μια πολύ πυκνή εβδομάδα και αυτό εξηγεί την απουσία πολλών μελών, αλλά θα ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία θα μας πείτε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας τη δημοσίευση του ΩΣΑ για θέματα μετανάστευσης. Θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να σας παρουσιάσω μια επισκόρπηση αυτής ε, της ε, έκθεσης των 400 τόσων σελίδων σε 12 περίπου λεπτά. Ας μου επιτρέψετε λοιπόν πρώτα να υπογραμμίσω τα βασικά μηνύματα τα οποία ε, βγαίνουν από την ανακοίνωση αυτή. Η μετανάστευση σύμφωνα με τον ΩΣΑ είναι στο υψηλότατο επίπεδο εδώ και δεκαετίες παρά μια μικρή μείωση που σημειώθηκε το 2017. Δεύτερον, ε, το, οι ισροές ετούντων άσυλο και προσφύγων φτάνει σε ένα νέο επίπεδο κανονικότητας. Έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο στα πλαίσια αυτής της έκθεσης σχετικά με τις ε, εξελισσόμενες αυτή τη φάση ροές μεταναστευτικές και προσφυγικές ε, παντού στην Ευρώπη θα είναι μεν χαμηλού ποσοτικού επίπεδου αλλά θα έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να δούμε ακριβώς και την επίπτωση που έχουν στις τοπικές αγορές εργασίας ε, ε, φαινόμενα όπως η παρουσία παράνομων μεταναστών. Ξεκινάμε λοιπόν. με τα στατιστικά στοιχεία α, να έχουν υποστεί επεξεργασία ή ασδήποτε μορφή επεξεργασία. Βλέπουμε συνολικά στις χώρες του ΩΣΑ 5 εκατομμύρια, το 40% έρχονται για λόγους οικογενειακούς, το 20% για ανθρωπιστικούς λόγους. 1,4 προέρχονται από τρίτες χώρες, ε, περίπου 300.000 περισσότεροι συνολικά από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε περίπου το ίδιο ποσοστό. Υπάρχει και το θέμα της εσωτερικής μετακίνησης των πολιτών. Αντίστοιχα έχουμε τα ίδια ποσοστά αν θέλετε μετακινούμενων εργαζομένων από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχουν βέβαια τεράστιες διαφορές ανάλογα με τη χώρα. Σε κάποιες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ε, Λετωνία, η Σλοβακία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε 3,4 ε, στο Λουξεμβούργο πάνω από το 2% στην, στην Ελβετία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από τις εσωτερικές μετακινήσεις κάτι πάνω από το 4% σε ετήσια βάση. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι η προσωρινή μετανάστευση για λόγους εργασίας είναι σε αύξηση εκτός από την κατηγορία των αποσπάσεων στο εσωτερικό ομίλων επιχειρήσεων. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι αυξήθηκαν το 16 κατά 30% λόγω μίας χώρας συγκεκριμένη της Πολωνίας. Για πρώτη φορά ε, βλέπουμε στα πλαίσια αυτής της κατανομής να λάβουμε υπόψη μας και στοιχεία για τους προσωρινούς εργαζόμενους, εποχιακούς εργαζόμενους στις χώρες του ΩΣΑ, ε, ε, όπως είπαμε 4 εκατομμύρια και η πρώτη χώρα ε, η οποία υποδέχεται προσωρινούς μετανάστες είναι η Πολωνία πριν από τις Ηνωμένε Πολιτείε και πριν από τη Γερμανία. Όλοι ίσως γνωρίζουν την κατάσταση στην Πολωνία και νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε για το 2017 θα έχουν ακόμα και ψηλότερα ποσοστά εποχιακών εργαζομένων. Σχετικά τώρα με, τους, ε, ε, με αυτούς που ζητούν άσυλο και τις πρόσφατες αφήξεις. Θυμάστε τι είχε συμβεί το 2016. 4 εκατομμύρια κόσμος ε, είχαν κάνει αίτηση για χορήγηση ασύλου ανάμεσα στο 11 και στο 14 στις χώρες του όσα 1,6 εκατομμύρια έτυχαν ε, διεθνούς προστασίας αλλά τους αριθμούς αυτούς ε, πρέπει να τους δούμε πολύ προσεκτικά για χώρες όπως ε, ο Λίβανος, η Συρία, η Τουρκία κτλ. Ξέρουμε επίσης τι συμβαίνει στο σύνολο της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού που έχουμε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ευρώπη λοιπόν έχει με αρκετά μεγάλους αριθμούς αλλά προφανώς βλέπετε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα είναι περίπου παρόμοια. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία έχουμε παρά τις ε, συνεχιζόμενες εντάσεις η Ευρώπη δεν έχει να αντιμετωπίσει στην παρούσα φάση μεταναστευτική κρίση. Από το 2018 η Ισπανία έχει ε, σημειώσει 50% περισσότερες αφήξεις από την Ιταλία και την Ελλάδα μαζί. Παρόλα αυτά είμαστε 10 φορές χαμηλότερα από ότι το 2015-16. Το θέμα τίθεται βέβαια σε πολιτικό επίπεδο. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι ε, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ για τις εγκαταστάσεις ε, προσφύγων στα πλαίσια των χωρών όσα μετά από την κορυφή των 120.000 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016, το 2017 φτάσαμε στις 60.000 παρά το ότι ένας αριθμός μετεγκαταστάσεων προς την Ευρώπη έχει κατά κάποιο τρόπο αυξηθεί. Επιμέρους λοιπόν αυξήσεις ειδικών κατηγοριών, συνολικά ο αριθμός όμως των μεταναστών έχει μειωθεί ε, από το 16. Μία ερώτηση η οποία έχει τεθεί είναι η επιπτώσει στην αγορά εργασίας. Στην επόμενη διαφάνεια και στην μεθεπόμενη διαφάνεια θα δούμε κάποια από τα στοιχεία. Το 2018 προσπαθήσαμε στην έκθεσή μας να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτές μέχρι το 2020 επί τη βάση διαφορετικών σενάριων. Το ένα σενάριο λέγει ότι οι ροές θα συνεχίσουν σε σχέση με αυτά τα οποία παρατηρήσαμε το 2011-2013. Ένα άλλο σενάριο θεωρεί ότι θα παραμείνουμε στην, ε, στο επίπεδο του 2017. Αυτό το οποίο φαίνεται εδώ είναι ότι μέχρι το 2020 θα έχει αυξηθεί το εργατικό δυναμικό λιγότερο από 0,23%. Δεν μιλάμε για κανένα σοκ σε επίπεδο αριθμών δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να ανησυχήσει την αγορά εργασίας, ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ελλάδα ή η Σουηδία, ε, μιλάμε για επιρροή 0,6 μέχρι 0,8 του εργατικού δυναμικού. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να διαταράξει δηλαδή τις ισορροπίες και τα ποσοστά και βλέπουμε ότι οι προβλέψεις μας μέχρι το 2020 σε όλους τους τομείς βλέπουν ε, πάρα πολύ χαμηλές επιπτώσεις. Πέραν τούτου και περνάω στην επόμενη διαφάνεια, δεν μπορείτε να το δείτε ίσως πάρα πολύ καλά από εκεί που είστε. Δείχνει εδώ ότι για κάποιες ειδικέ κατηγορίες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Αυτό ισχύει για άνδρες χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου από 18 μέχρι 34 ετών. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν δηλαδή στην Ευρώπη ε, ανήκουν ιδιαίτερα σε τέτοιες κατηγορίες και μπορεί να επηρεάσουν κατά 15% τις αντίστοιχες κατηγορίες εργατικού δυναμικού τη συγκεκριμένη επαναλαμβάνω κατηγορίας. Βέβαια αυτή η ομάδα ποσοστιαία δεν είναι και αυτή πάρα πολύ υψηλή ακόμα και το κακό σενάριο για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και λόγω και του ανταγωνισμού υπάρχει στην ουσία μια σύγχυση από πλευράς του κοινού, η εικόνα την οποία έχει το κοινό είναι ε, πολύ πιο ε, ευρεία σχετικά με το πραγματικό μέγεθος του φαινομένου. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά για νέους άνδρες οι οποίοι έχουν ε, χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Ένα τελευταίο τώρα να πω στα επόμενα δύο λεπτά αναφέρεται στην παράνομη χρήση ξένων εργαζομένων. Ήδη από το 2015 είχαμε πει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ. Υπήρξαν πάρα πολλά μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και πρόσφατα υπάρχουν κάποια φαινόμενα που ενισχύουν δυστυχώς το φαινόμενο. Καταρχάς, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 2008-2009 Πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες είχαν χάσει τις θέσεις απασχόλησής τους. Δεν ήσαν παράνομοι τότε, αλλά χάνοντας τη θέση απασχόλησής τους, στην ουσία μετετράπησαν σε παράνομους. Αλλά, όπως βλέπετε, υπάρχουν και αυξανόμενοι αριθμοί μεταναστών στους οποίους δεν δίδεται το καθεστώς του ασύλου και αυτό τους καθιστά και αυτούς παράτυπους μετανάστες Συνολικά η κατηγορία αυτή για το σύνολο της Ένωσης ποικίλει από 900.000 μέχρι 1,1 εκατομμύρια. Η επόμενη διαφάνεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε υπάρχει η κατηγορία η οποία δεν είναι συμβατή με συγκεκριμένους κανόνες ή με το σύνολο των κανόνων. Γενικά είναι ένα πολυδιασπασμένο αλλά και περίπλοκο φαινόμενο μπορεί να συνδέεται με τους λόγους τους οποίους προανέφερα. Ε, υπάρχουν κατηγορίες ε, στους οποίους οι άδειε εργασίας τις οποίες κατήχαν νόμιμα έχουν ε, πλέον λήξει οπότε περνούν σε διαφορετική κατηγορία πολλές φορές εργάζονται στον ανεπίσημο θα λέγαμε τομέα οπότε δύσκολα θα μπορούσαν να βγάλουν χαρτιά. Στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, το 3,5 του πληθυσμού ε, είναι πρόσφυγες και μετανάστες αλλά στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βγάλουμε τέτοια στοιχεία αλλά σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερο το συγκεκριμένο φαινόμενο αυτό και περιορίζεται σε τομείς όπως η γεωργία, οι οικοδομές και η ε, βοήθεια στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά βασική, όλα... λόγη για την απασχόληση των ε, λαδαπών εργαζόμενων. Υπάρχει ε, αναντιστοιχία ανάμεσα στη ζήτηση για ε, χειρονακτικές ε, εργασίες ή εργασίες ε, χαμηλής εκπαίδευση. Ε, Επειδή υπάρχει κενό ανάμεσα στην, στα συνέπειες στις διοικητικές, διοικητικούς κανόνες και πλαίσια που μπορεί να προκαλέσουν παρατυπίες και τέλος είναι χαμηλά τα κίνητρα για τους, για τους εργοδότες να προσλαμβάνουν νόμιμους εργαζόμενους λόγω της ιχνής ε, επιβολής της ε, σχετικής νομοθεσίας στον χώρο εργασίας. Ποιες είναι τώρα οι απαντήσεις που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ε, φυσικά η ενημέρωση και η επαλήθευση να γίνονται προσπάθειες ε, με συγκεκριμένα μέσα, έλεγχος και επιβολή. Οι περισσότερες χώρες στοχεύουν ειδικού τομεί με επιθεωρήσεις εργασίας μαζί με τυχαίους ευρύτερους ελέγχους. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα μέσα, τα οποία για την ώρα είναι λιγοστά, κυρώσεις και ποινές Ε, είναι πολύ διαφορετικές οι προσεγγίσεις, αλλά τελικά φαίνεται να ε, κυμαίνεται τόσο η αποδοτικότητα και όσο και η αποτελεσματικότητα των ε, ελέγχων αυτών για να αλλάξουν την στάση των εργοδοτών. Η πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης ήταν πολλά μέτρα μέσα, ε, μέτρα μάλλον για την αγορά εργασίας, ε, μέτρα για την μετανάστευση και ε, τρόποι για να επιβληθούν τα ισχύοντα μέτρα και σαφώς σε πλαίσιο ευρωπαϊκό η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης δίνει πολλές ευκαιρίες για να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτού του είδους ε, η κατάσταση πέμπτη απόγευμα όπου πολλά μέλη ε, λείπουν, ε, να ξέρετε ότι οι συνεδριάσεις μας αναμετωδίδονται στο διαδίκτυο ε, και μπορεί κανείς να παρακολουθεί ακριβώς τι γίνεται από αλλού ε, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και εγώ έχω διάφορες ερωτήσεις από ό,τι βλέπω και η κυρία Γκόμες. Η δική μου ερώτηση για το κατά πόσο καταγράφονται λοιπόν όλα αυτά είναι καταρχάς ε, ότι τώρα είμαστε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου η οικονομική μετανάστευση παρουσιάζεται με αρνητικό πρόσημο. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες χώρες. Μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτού του είδους η ασθένεια είναι διαδεδομένη. Ε, εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τις οικονομικές προβλέψεις και όσον αφορά τη μετανάστευση, γενικό μου ερώτημα είναι ε, ποιες είναι οι προβλέψεις, γιατί η οικονομία έχει σημασία. Ποιες είναι οι προβλέψεις για το άσυλο και την μετανάστευση. Και πώς βρίσκεται, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο βλέπετε να υπάρχει ένα θέμα ότι δεν εξετάζονται σοβαρά οι προβλέψεις. Έπειτα, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία, όπου γνωρίζουμε ποια είναι η τάση. Ας πούμε, ο αριθμός των διελεύσεων ε, στην Μεσόγειο έχει μειωθεί και αυτό Ε, είναι κάτι που το αναμένουμε όταν βλέπουμε ότι οι αιτήσει για χώρες του ΩΣΑ έχουν μειωθεί. Ο ΩΣΑ όμως θεωρείται πολύ αξιόπιστος οργανισμός, οπότε βρίσκεται ότι όταν μιλάτε για αυτά τα θέματα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουν ότι τα νούμερα μειώνονται Οι αιτήσει δηλαδή ασύλου μειώνονται και μειώνονται ακόμη και περισσότερο τώρα. Υπάρχει καθόλου επιμονή στο να το δείξετε αυτό και να το αποδείξετε. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που τώρα καλύπτουμε είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας, η ολοκλήρωση. Παλιότερα το έκανε αυτό η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Επασχόλησης, αλλά τώρα έχει περιέλθει στις δικές μας αρμοδιότητες αυτό το θέμα. αυτό που λέτε για κάλυψη της αγοράς εργασίας από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τα νούμερα πιστεύετε ότι προχωρούν στην σωστή κατεύθυνση, δηλαδή βλέπουμε καλύτερα νούμερα Ε, για Αφρικανούς ή σε σχέση με Ασιάτες ας πούμε ή άλλους αυξάνονται. Οπότε δηλαδή βλέπετε να διαγράφεται στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν διάκριση. Ε, εντάξει, δεν υπερβάλλουμε με τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως βελτιώνονται τα πράγματα. Με αυτό τώρα το νούμερα που εσείς ε, παρουσιάζεται, βλέπετε να υπάρχει κάποια πρόοδος, οι κυβερνήσεις τα χρησιμοποιούν, οι ΜΚΟ τα χρησιμοποιούν, οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ή τα αγνοούν. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται. Γιατί είναι νούμερα που μετρώνται σε πολιτικώς ευαίσθητους τομείς. και λένε διηγούνται μια σχετικά θετική ιστορία. Ότι δηλαδή βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά οι πολιτικές αντιδράσεις ε, κατά των μεταναστών είναι χειρότερες, ενώ δημογραφικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ωστόσο η αποδοχή των μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι αρνητική. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης λοιπόν είναι οι ερωτήσεις μου και πάλι ως προς τον ΩΣΑ για το θέμα της αξιοπιστίας κάνετε εσείς προβλέψεις για τον οικονομικό τομέα Για την νόμιμη μετανάστευση, ελπίζω πως η Κομισιόν δεν θα εγκαταλείψει αυτή την πρόθεση για νόμιμη μετανάστευση και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Πρέπει ωστόσο να έχουμε αξιόπιστες στατιστικές, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε σωστά. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε ε, εργαλεία νόμιμης μετανάστευσης τα οποία να λειτουργούν εύρυθμα και σωστά ε, πρέπει να εξετάσουμε τέτοιου είδους ε, εκθέσεις. Ελπίζουμε και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και νέα για την νόμιμη μετανάστευση. Θα δούμε τι θα γίνει με εκείνες τις προτάσεις. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ και με ενδιαφέρει η εμπειρία σας πίσω από όλα αυτά τα νούμερα. Άννα, έχεις ερωτήσεις για τον ΟΣΑ, για την μετανάστευση. Όχι. Μάλιστα, εγώ σας έβαλα όλες τις ερωτήσεις, αλλά πολύ με ενδιαφέρει το θέμα, οπότε... Και είμαι ευγνώμων που ήρθατε και μας κάνατε αυτή την παρουσίαση. Παρακαλώ λοιπόν για πείτε μου τι πιστεύετε για όλα αυτά που σας ρώτησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την ευκαιρία που μου δίνετε και πάλι γιατί έτσι έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις πληροφορίες. είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τα κοινοβούλια ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι αλλαγές και η εξέλιξη της κατάστασης. Όπως την παρουσιάζουν οι στατιστικές, θα έλεγα, σε σχέση με την ερώτησή σας δηλαδή για το βαθμό στον οποίο τα νούμερα που συζητάμε είναι χρήσιμα και εισακούγονται, αυτό εξαρτάται πιστεύω πολύ από τη δυνατότητα που έχει κανείς να κατανοήσει τι δημιουργεί την αποσύνδεση ανάμεσα στη δημόσια, στην κοινή γνώμη και τους εμπειρογνώμονες ή και τις στατιστικές. Και μέρος όλων αυτών πιστεύω ε, οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να ε, ξεπεράσουμε ε, αυτά τα θέσματα. Τα λέμε δηλαδή ότι η, ε, η μετανάστευση θα αυξήσει το εργατικό δυναμικό, αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τι θα μπει στην τσέπη τους. Και όσον αφορά τους μετανάστες, ε, το νούμερο μπορεί να είναι μικρό, αλλά μπορεί να υπάρξει συγκέντρωση σε κάποιες ε, περιοχές, σε, κάποιες, ε, σε κάποια μέρη. Είναι σημαντικό λοιπόν στην ανάλυση να μην, να μην αγνοούμε αυτή την ανησυχία, να το εισακούσουμε και να ξεπερνάμε τους μέσους όρους, να δίνουμε τους μέσους όρους, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα σημεία όπου προκύπτουν οι ανησυχίες. Και αυτό κάνουμε και σε αυτή την έκθεση γενικά. Όταν πρόκειται για συγκεκριμένες ομάδες, δηλαδή εγκατάλειψη του σχολείου, νέοι άνδρες, που ήδη δημιουργούν πολλά προβλήματα, τότε εκεί τα νούμερα μπορεί να παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Και εκεί πιστεύουμε ότι θα μπορούσε αυτό να καθοδηγήσει την αντίληψη περί μέσου όρου αντικτύπου. Επίσης σε, σε αυτή τη δημοσίευση αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εισακούσουμε τις ανησυχίες. Το να συζητάμε για την παράνομη μετανάστευση είναι λάθος. Γιατί αν θέλουμε να εξηγήσουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε κανόνες, να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, και να μπορεί να παραμείνει, να έχουμε, θα πρέπει να έχουμε εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο έκανε μια έρευνα με την ερώτηση «Πιστεύετε ότι περισσότεροι μετανάστες ε, είναι νόμιμοι ή παράνομοι» Το 40% των Ευρωπαίων έλεγαν ότι υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που είχαν τακτοποιημένη την κατάστασή τους και αυτό ήταν λάθος. Αλλά αυτή ήταν μια αίσθηση που επικρατούσε. Γι' αυτό και το βλέπουμε, το εξετάζουμε αυτό, παρά το ότι έχουμε δυσκολίες όσον αφορά τα δεδομένα, ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τόσο δύσκολα ζητήματα και να βρούμε αποδείξεις ε, που βάζουν τα πράγματα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι ένα θέμα, όπως είπαμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έγκυρη άδεια παραμονής, αλλά ζουν και εργάζονται άτυπα. Άλλοι που ε, δεν έχουν ε, άδεια παραμονής, αλλά είναι δηλωμένοι από τον, απασχολ, από τον εργοδότη τους. Είναι δηλαδή ανάμεκτη κατάσταση. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα αυτά. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε λοιπόν Όσον αφορά τα νούμερα, και είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να διοχετευθούν στο ευρύ κοινό, αλλά προσπαθώντας να εισακούσουμε τις ανησυχίες και να ακολουθήσουμε ε, μια πορεία πέρα από τους μέσους όρους, ε, προσπαθούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο ΣΑ κάνει κάποιες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη και λέει ότι θα γίνει το τάδε το δεινά. Θα, θα ήταν καλό ίσως να είχαμε κάτι παρόμοιο και για την μετανάστευση. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά σας και πολύ αξιόπιστη. Ε, και γι' αυτό ήμασταν ευτυχεί που, είχα, που σας είχαμε σήμερα εδώ, ακόμα και αν ανταλλάξαμε απόψεις σε ένα, ένα έτσι πιο χαλαρό ρυθμό, καθότι είναι πέμπτη απόγευμα, αλλά όπως σας είπα, οι συνεδριάσεις μας αναμεταδίδονται στο διαδίκτυο και όποιο θέλει μπορεί να τις παρακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ο Πρόεδρος, συνεχίζουμε συνάδελφοι, είμαστε κάπως νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ο κύριος Γκρέγορ είναι παρόν. and we can then uh, we can start the new point a wee bit earlier. Yeah, Ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν επιτρέπετε να αρχίσουμε με το θέμα 14 για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόκειται για παρουσίαση του μέλους του παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριο Γκρεγόρ. ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Καλώς ορίσατε. Είστε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ποιότητας Ελέγχων. Ένα από τα αντικείμενά σας είναι ο έλεγχος της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και είναι πολύ ενδιαφέρον που το ελεγκτικό συνέδριο το εξετάζει. Μπορώ να σας δώσω 15 λεπτά. Σας ε, επισημαίνω ότι ναι μεν είναι λίγα μέλη του Κοινοβουλίου παρόντα, ωστόσο μεταδίδεται η ομιλία σας από το διαδίκτυο σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πρώτα για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τον έλεγχο της ριζοσπαστικοποίησης. Είχαμε ήδη συναντηθεί στη πρώτη των θερινών διακοπών με σε κοινή συνεδρίαση δύο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών μιλούμε για θέματα μετανάστευσης και ενδεχομένως ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να ακολουθεί. Ας έλθουμε τις διαφάνειες της ε, παρουσιάσεως που έχω συντάξει ειδικά για τη σημερινή σας συνεδρίαση. Καλύπτω πέντε τομείς, δηλαδή ποια είναι η προσέγγιση ελέγχου και στα δύο τελευταία που βλέπετε στην οθόνη σας είναι οι συμπεράσματα και συστάσεις. ασφάλεια και αγώνας κατά της δημοκρατίας είναι ζήτημα αρμοδιότητας των χωρών μελών. Εντός δε των χωρών μελών αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση διότι η κατάσταση και οι προκλήσεις εξαρτώνται πολύ από τα τοπικά δεδομένα. Και η προσέγγιση αυτή είναι σημαντική. Από την σκοπιά αυτή, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προσφέρει στήριξη στι χώρε μέλη, στι προσπάθειέ του για την διασφάλιση τη εφαρμογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών με ποιότητα και εγκαίρω. Στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε τώρα σας εξηγώ γιατί αποφασίσαμε να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε τον τομέα αυτό το 2005 εγκρίθηκε αντιτρομοκρατική πολιτική, χωρισμένη σε διάφορους πυλώνες, πρόληψη, αντίδραση, καταστολή, αντιμετώπιση της ροσβαστικοποίησης, ισχυρότερη ασφάλεια συνόρων, διαρεύνηση τρομοκρατίας και αντιμετώπιση συνεπειών επιθέσεων. Ο έλεγχός μας αναφέρεται στον πρώτο πυλώνα, στην πρόληψη, με διερεύνηση των αιτίων της ρίζοσπαστικοποίησης που συνδέεται με την τρομοκρατία. Επιλέξαμε να ρίξουμε τα φώτα μας εκεί, διότι σε πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτές έγιναν από ριζοσπαστικοποιημένους Ευρωπαίους πολίτες. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων παραγόντων, κοινωνικών, παραγόντων όπως περιθωριοποίηση και αποκλεισμό επίσης ιδεολογική έλξη με τα αφηγήματα των στρατολογητών από την πλευρά ε, αυτών που θέλουν να προχωρήσουν σε παράνομες πράξεις. Σημαντική και πολυσχηρής πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ριζοσπαστικοποίηση με δράση σε διάφορους τομείς πολιτικής, χρησιμοποιώντας και κονδύλια που διαχειρίζονται οκτώ διαφορετικές γενικές διευθύνσεις με μία ενιαία εντολή. Εσωτερική ασφάλεια, ορίζον 2020, αυτά είναι τα διάφορα κονδύλια, τα μία τα οποία χρησιμοποιούνται έρασμος συν και τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ποιες είναι οι ερωτήσεις που θέσαμε εμείς. Ρωτήσαμε εάν η στήριξη προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή εκεί όπου τη, όπου τη χρειάζονται οι χώρες μέλη, εάν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σχεδιασμένες ώστε να αποφέρουν ωφέλη στις χώρες μέλη, ώστε να είναι υποφελής η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια το θέμα είναι τόσο σημαντικό και οριζόντιο, ώστε χρειάζεται συντονισμός των διαφόρων δράσεων και πηγών χρηματοδότησης για να αναπτυχθούν οι περισσότερες δυνατές συνέργειες. Ερευνήσαμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προσπάθεια για να διασπείρει τα συμπεράσματα και πορίσματα των δράσεων αυτών, αν μετρά την αποτελεσματικότητα της στήριξης που προσφέρει. Στην επόμενη διαφάνεια εξηγώ πώς διεξήχθη ο έλεγχος. Κάθε έλεγχος αρχίζει με έλεγχο της τεκμηρίωσης. Κάναμε επίσης συνεντεύξεις, συναντήσεις δηλαδή, με μέλη του προσωπικού της Κομισιόν. Έχουμε τα κέντρα υπεροχής στο Άμστερνταμ και τα γραφεία της Ευρωπόλ στην Χάγη, όπου ήρθαμε σε επαφή με τους αρμοδίους. Συναντηθήκαμε με αρμοδίους σε όλες τις χώρες μέλη. Δεκαπέντε χώρες μέλη απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας, 54% δηλαδή. Επισκεφθήκαμε δε τις εθνικές αρχές σε Γαλλία και Βέλγιο για να συζητήσουμε μαζί τους ε, τι σημασία αποδίδουν στη στήριξη που τους προσφέρει η Επιτροπή. Αποτελέσματα. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στην πρώτη μας ερώτηση, εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει κατάλληλη στήριξη στις χώρες μέλη. Γενικά το συμπέρασμα είναι μάλλον θετικό. Η συνολική στήριξη που δίνεται είναι καλά σχεδιασμένη και επαρκής. Αντιμετωπίζει σωστά τις ανάγκες των χωρών με κάποιες εξαιρέσεις, αποφέρει ωφέλη στις χώρες μέλη από τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει τις ανάγκες των χωρών στην γνώση περί ριζοσπαστικοποίησης με έρευνα, με ε, διάδοση των πορισμάτων, αντιμετώπιση της ριζοσπαστικής προπαγάνδας μέσω του διαδικτύου, με ε, μηχανισμούς του ΣΥΝ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διευκολύνσεις επαφών μέσω του συστήματος προφοριών Schengen και τέλος αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, προγράμματα που ε, υποστηρίζει χρηματοδοτικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το έργο αυτό της Επιτροπής είναι καλά σχεδιασμένο, βρήκαμε. με το Euro Internet Forum και με το δίκτυο ε, στρατηγικών επικοινωνιών. Διαπιστώσαμε ότι αυτά γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο και καλύτερα από ό,τι θα γίνονταν από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Τώρα για την απάντηση που δώσαμε στη δεύτερη ερώτησή μας. Αν είναι επαρκής ο συντονισμός για να υπάρξουν συνέργειες. Βρήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφυριλατεί συνέργειες, υπάρχουν όμως ορισμένοι τομείς όπου μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός. Υπάρχουν και συνέργειες μεταξύ ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα για την αξιολόγηση των δράσεων κατά της ριζοσπαστικοποίησης. και με χρήματα του Ερασμοσύμ. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, υπάρχουν ελλείψεις στον συντονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει, για παράδειγμα, πλήρη εποπτεία όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δε RAN δεν χρησιμοποιείται για, στο πλήρες δυναμικό του. Από τα 16 προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο σχετικός συντονισμός γίνεται μόνο για 7. Στην τρίτη μας ερώτηση, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει κατάλληλο πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεών της, βρήκαμε ότι το δίκτυο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένο. Το εξετάσαμε αυτό σε δύο επίπεδα συνολικής πολιτικής και επιμέρους δράσεων Βέβαια οφείλω να πω ότι για μια τέτοια σημαντική πολιτική που πρέπει να αναπτυχθεί και με ταχύτητα για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές, νομίζω είναι κατανοητό ότι κάπως υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Αλλά πρόκειται για ένα τομέα τον οποίο οφείλει να εξετάσει το ελεγκτικό συνέδριο. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπω για παράδειγμα την Internet Refer Unit της Ευρωπόλ που αναφέρεται σε παρόχους υπηρεσιών όπως Facebook, Twitter κλπ. Και αναφέρει σε αυτές τις πλατφόρμες ε, ιστοσελίδες τρομοκρατικού περιεχομένου με το αίτημα να αφαιρεθούν. Και βλέπετε εδώ τους αριθμούς των ε, ιστοσελίδων που αφαιρέθηκαν με ένα συνολικό ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 80%. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για το η τρομοκρατική παραπαγάνδα παραμένει στο διαδίκτυο. Και υπάρχει μέγας κίνδυνος η προπαγάνδα που έχει αφαιρεθεί να αναρτηθεί κάπου αλλού, σε άλλο σημείο του διαδικτύου. Να έρθω στις συστάσεις μας. Στην έκθεσή μας κάνουμε τρεις συστάσεις. Η πρώτη μας σύσταση είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός δράσεων κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Βρήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίσει τις δράσεις της και τις βασικές συνεργές, αλλά υπάρχουν δύο τομείς όπου αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχει και κατάλογος δράσεων κατά της ριζοσπαστικοποίησης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το εθνικό επίπεδο και συστήνουμε επίσης να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το δίκτυο RAN, R-A-N Στην δεύτερη σύστασή μας προτείνουμε να συσταθεί η πρακτική στήριξη σε αυτούς που ασχολούνται στην πράξη με την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, να ακολουθηθεί μια λογική Βεβαίως υπάρχουν και τοπικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να αξιολογηθεί η τελική επιτυχία των δράσεων. Τέλος, η τρίτη σύστασή μας αναφέρεται στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τόνισα όμως και προηγουμένως ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι θα υπάρχει κάποια χρονική υστέρηση στο θέμα αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Γκρεγόρ. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεμελιωτών Ελευθεριών κατά τις 4. Κάτι τέτοιο θα ήταν καλό. Έχουμε κοντά μας τις ε, κυρίες Τσινίτσι ε, και Στίβενς διότι είχαμε και το θέμα του κόστους της μη Ευρώπης στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί και από δημοσιονομική σκοπιά. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, τα ίδια προσπαθεί να κάνει και η Επιτροπή ΤΕΡ, που είναι η Επιτροπή για την ε, Διερεύνηση της Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας. Βέβαια δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρεκόρ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κίνιτσι. Και θα ακούσουμε βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Κλόντ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ομιλητή για την παρουσίαση την οποία μας έκανε. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο, ίσως να είναι, ε, θα έλεγα, το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης ε, πολλές είναι οι αιτίε οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν μερικές φορές νεότατους ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Τους ευχαριστώ λοιπόν για τη σύνθεση την οποία μας έκανε, για την έκθεση. Υπάρχουν ε, θα έλεγα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν τη σημασία που έχει συνολικά η έκθεση, η στήριξη είναι απαραίτητη από πλευρά των κρατών μελών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς αναφερθήκατε στα ταμεία που χρηματοδοτούν τα προγράμματα. Θα ήθελα να ζητήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει ένα πλήρη κατάλογο των δράσεων που έχουν αναλυφθεί σε κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερη για τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορέσει να διευκολύνει αυτό το οποίο είπατε, την διάδοση δηλαδή των σωστών αποτελεσμάτων και των χρήσιμων αμοιβαία πρακτικών. Στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχουν των ειδικών ε, εξουσιών στον τομέα της ασφαλείας τους. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μωράης, είμαι εδώ, είμαι στη Λίμπε, είμαι στην Τέβε και προσπαθώ να ακολουθήσω τα θέματα αυτά από διαφορετικές προοπτικές. Μια άλλη πλευρά είναι ότι η έκθεση αυτή αποδεικνύει το πώς ε, οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας δεν έχουν γίνει αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του ουράν και να ανταλλάξουμε τις λεγόμενες χρηστές πρακτικές. Λείπει λοιπόν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιου είδους δράσεων. Οι δείκτες οι οποίοι υπάρχουν είναι επαρκείς, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τον Επίτροπο Κίνγκα. Είναι το θέμα της απομάκρυνσης από το διαδίκτυο των μηνυμάτων με τρομοκρατικό περιεχόμενο. Αναφερθήκατε και σε αυτό. Ε, μπορεί να συμβεί μερικές φορές περιεχόμενα τα οποία αναγνωρίζονται από την ε, μονάδα ίντερνετ της Europol να αποσυρθούν από ένα site. Υπάρχει ο κίνδυνος όμως να δημοσιευθούν σε ένα άλλο site. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι μερικές φορές θα έχουμε την, σε μερικές μέρες συγγνώμη, θα έχουμε την πλήρη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια μέτρα τα οποία να αποτρέψουν τον κίνδυνο αυτό, να απομακρύνουν τον κίνδυνο αυτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε λοιπόν εσείς να σχολιάσετε λίγο αυτά τα οποία σας είπα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας η οποία ήταν πληρέστατη. Ευχαριστώ πολύ Κατερίνα. Και έτσι μπορούμε να είμαστε και να ανταποκριθούμε σωστά σε αυτό το σημαντικό έργο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Η Κομισιόν ήθελε να πάρει το λόγο. Ο Ολιβιέ ε, είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα είμαι σύντομος. Είχα την ευκαιρία να πω δύο λόγια στην Επιτροπή Κοντ και Τέρα και είμαι ευτυχής που μπόρεσα να είμαι σήμερα εδώ γιατί, γιατί η έκθεση είναι πολύ καλή η έκθεση ήταν επίσης έγκαιρη γιατί μπορεί να ενσωματωθεί στη συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επίπεδου που συστήσαμε πριν από 1,5 χρόνο για την ε, ε, ρεζοσπαστικοποίηση και ε, θα είναι και κομμάτι των δράσεων που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Σύντομα να σας πω ότι έχουμε ήδη κάνει όταν δούμε το τρία σύνολα συστάσεων για τον συντονισμό. Έχουμε αντιμετωπίσει τον εσωτερικό συντονισμό ε, σε, με, την σύσταση της Task Force όπου συμμετέχουν διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν που παίζουν ρόλο και δι, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ρίζοσπαστικοποίησης. Επίσης, καταφέραμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στους ε, ε, επιτόπου εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα στο πλαίσιο του δικτύου ΡΑΝ, αλλά και τους ηθήνοντες για την πολιτική, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στις διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη μεγιστοποίηση της ε, χρήσης των διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων όχι μόνο πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί και να δώσουμε αποτελέσματα, αλλά θα είδατε και ότι πολλά από αυτά έχουν ε, παρουσιαστεί εδώ στην ε, ΛΥΜΠΕ, τα, τα εγχειρίδια για τα παιδιά, για τις φυλακές, ε, για το σύνολο συζητήσεων και συστάσεων σε αυτό το τομέα που παραμένει εξαιρετικά δύσκολος, όπως είπατε, ε, πρόεδρε, στην αντιμετώπιση του. Ε, έχουμε και μια ενδιάμεση εξπόστα αξιολόγηση την οποία θα κάνουμε, θα τη δούμε με τα διάφορα μέσα που έχουμε στην ε, ε, διάθεσή μας ε, να φτιάξουμε και δείκτες προσπαθούμε που είναι δύσκολο να το επιτύχουμε γιατί τα αποτελέσματα συχνά δεν είναι ε, αξιόπιστα, δεν είναι πάντα ακριβή και επίσης το υλικό από το ίντερνετ που πρέπει να αφαιρεθεί από το ίντερνετ και μετά ξανά εμφανίζεται πολύ συχνά σε άλλες πλατφόρμες. Μετά έχουμε ε, αυτό που μεταφράζεται σε μια αυτόματη αφαίρεση του συγκεκριμένου υλικού από όλες τις διάφορες πλατφόρμες που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Θα είναι ένα κομμάτι της πρότασης που θα ανακαλύψουμε την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των εταιριών ε, ίντερνετ με τις οποίες συνεργαζόμαστε ώστε να δουλέψουμε για αυτά, με αυτές τις πρωτοβουλίες και τέλος ε, έχουμε θεσπίσει ένα συστηματική, μια συστηματική αξιολόγηση κάθε φορά που σταματά μια δραστηριότητα έχουμε μια αξιολόγηση ε, των δραστηριοτήτων. Τα μέτρα αυτά λοιπόν έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τον εστιασμό σε όσους φύγουν από, φεύγουν από την Ευρώπη για να πάνε σε κάποιο πεδίο μάχηση και αντίστροφα και πιο σημαντικά αυτούς που ενεργούν ε, στη χώρα τους. Να αποφύγουμε δηλαδή την ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων στις χώρες μας. Να αποφύγουμε τρομοκρατικές επιθέσεις εδώ. Η φυλακή ε, προσπαθούμε να, να κινηθούμε περισσότερο προς αποκατάσταση και προς την πρόληψη. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για αυτά τα πολύτιμα λεπτά. Έχουμε κάποια τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να κλείσουμε την συνεδρίαση σύντομα. Σας παρακαλώ λοιπόν να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ τέσσερα θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προωθήσουμε νομίζω σε, όλες, σε όλα τα κράτη-μέλη την πρωτοβουλία αυτή, γιατί δεν ε, συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη ενεργά. Για το περιεχόμενο στο ίντερνετ, εγώ προσωπικά πιστεύω πως είναι σχεδόν αδύνατη αποστολή, γιατί ε, Ακόμα και αν εξαφανιστεί από το ίντερνετ, μπορεί να, μπορεί να ξαναεμφανιστεί στο darknet ή σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Ο κίνδυνος υπάρχει πάντα. Ξέχασα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εξαιρετική συνεργασία στη διάρκεια της εκτέλεσης αυτού του ελέγχου. Θέλουμε λοιπόν ε, να σας πούμε ότι αργότερα φέτος θα παρουσιάσουμε ένα ενημερωτικό έγγραφο για την κυβερνοασφάλεια και μέσα στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σκοπεύουμε να συντάξουμε έκθεση για το κατά πόσο τα συστήματα της Ένωσης στηρίζουν τους συνοριακούς ελέγχους. Και εγώ και συνάδελφοι θα έρθουμε στις διάφορες επιτροπές για να σας ενημερώσουμε και για αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη, κυρία Στίβεν, είχατε ζητήσει το λόγο, αλλά δεν σας είδα. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα σύντομα. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας είδα. Ναι, αν θέλετε τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Ναι, πρόεδρε, είχα σηκώσει το, το, το, το, χέρι μου, αλλά μάλλον δεν με είδατε. Για το θέμα της τρομοκρατίας θα ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα υπάρχουν ε, μέθοδοι για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των ε, προγραμμάτων και δαπανώνται διάφορα εκατομμύρια για τα project αυτά κατά της ζωσπαστικοποίηση Λειτουργούν όμως πραγματικά, γιατί εδώ μιλάμε για κέντρα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Προβλέπονται ε, κριτήρια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών το project, αλλά... Εσείς τι πιστεύετε, είναι αποτελεσματικά. Thank you very Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που δεν σας έδωσα νωρίτερα το λόγο. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας ε, απαντήσετε με μία email για να τις δώσετε τις λεπτομέρειες ε, που μπορεί να έχετε συγκεντρώσει και απαντήσεις και να έρθετε μαζί της άμεσα σε διάλογο. Ναι, και είναι και για την Κορομισιόν η απάντηση αυτή, οπότε πρέπει να τα στείλουμε και στην Κομισιόν. Μάλιστα, θα σας, θα σας ζητήσω λοιπόν να απαντήσετε. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ήταν τελευταία μας, ε, ε, το τελευταίο μας σημείο. Ε, εάν δεν υπάρχουν κάτι στα διάφορα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάντα όλους όσοι μένετε μέχρι το τέλος της ε, ολοκλήρωσης δηλαδή της ημερησίας μας διάταξης, καθώς και το σκληρά εργαζόμενο προσωπικό μας. Ε, να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες μας, νομική υπηρεσία και όλους όσοι είστε εδώ. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο για όλους.